Καθίστε παρακαλώ. Σήμερα καλούμαστε να εκφραστούμε και για τη συνολική οικονομική και εμπορική συμφωνία με τον Καναδά. Ήταν μακρά η διαδικασία και γεμάτη εμπόδια. Πιστεύω ότι δηλώθηκε η αντίθετη θέση. Κοιτάξτε, εδώ είμαστε στο Κοινοβούλιο, πρέπει όλοι να σέβονται τους κανόνες. Πολλοί εκφράστηκαν κατά τη συμφωνία αυτή. Πολλοί πολίτες ε, διαδήλωσαν ε, εκτός αυτής της αιθούσης για να εκφράσουν τις ιδέες τους. Σημαντικό είναι να σεβόμαστε πάντα τους κανόνες και τις ιδέες των υπολείπων. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να είναι πρωταγωνιστής και εγώ δεσμεύομαι, το καθήκον μου είναι να δράσω έτσι ώστε οι αποφάσεις που λαμβάνονται από αυτό τον οίκο να επιτρέψει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής δραστηριότητας γιατί οι πολίτες που όλοι εκπροσωπούμε πρέπει να γνωρίζουν ότι οι εκπρόσωποι τους υπερασπίζουν τα συμφέροντά τους. Όπως συνήθως, εγώ δεν θα ψηφίσω, όχι γιατί δεν έχω φυσικά τις μου ιδέες, αλλά επειδή κατά την κρίση μου η θέση του Προέδρου θα πρέπει να είναι η θέση που υιοθετείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε μια τόσο σημαντική ψηφοφορία. Να πω κάτι θετικό. Στις 6 ε, Φεβρουαρίου η βασίλισσα, του, η βασίλισσα της Αγγλίας γιόρτασε τα 65 χρόνια βασιλεία τη, και ελπίζω ότι οι συνάδελφοι από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Κοινοπολιτεία και από τη Μάλτα και από την Κύπρο θα χαιρετήσουν μαζί μου αυτό το ευτυχές γεγονό. Bene. Onorevole Valenciano. Μάλιστα. Κύριε Βαλενσιάνο. Ε, Μόνο μία ερώτηση κύριε Πρόεδρε. Δεν κατάλαβα πολύ καλά. Μία ερώτηση. Θα ψηφίσουμε τώρα ή δεν θα ψηφίσουμε ποτέ. Εγώ ως πρόεδρος δεν θα ψηφίσω ποτέ όταν προεδρεύω. Γιατί πιστεύω ότι είναι μια δική μου προσωπική επιλογή. Μπορώ να το κάνω. Η θέση του Προέδρου θα πρέπει να είναι η θέση του Κοινοβουλίου. Έχω λάβει από το ΕΛΚ ένα αίτημα για ένα διορισμό σε μία αντιπροσωπεία που θα καταγραφεί στα πρακτικά της συνεδρίασης. Αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις μέχρι την οθέτηση των πρακτικών, αυτός ο διορισμός θα θεωρηθεί ότι εγκρίνεται. Αφορά την Κοινοβουλευτική Συνέλευση τη Εκπροσώπηση και Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριο Ρεντζέλ θα την καταστήσει τον κύριο Ρουάς.